η έκθεση του Κάρλος Κοέγιο σχετικά με την κυκλοφορία προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής. Περιμένουμε την κυρία Βάλστρομ να καθίσει. Welcome. Καλώς ορίσατε. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή μας, τον κύριο Κοέγιο, να μιλήσει για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε παράλογε περιπτώσεις όπως ένας φοιτητής ο οποίος παίρνει θεώρηση για να παρακολουθήσει ένα, κάποια μαθήματα στο Βέλγιο και δυστυχώ, δεν θα μπορεί να πάει στην Ολλανδία να σπουδάσει, ε, να εκμεταλλευτεί μια βιβλιοθήκη ή να πάει ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη γιατί ουσιαστικά είναι ε, φυλακισμένος στη χώρα αυτή. Μιλάμε λοιπόν για θεωρήσεις μακράς διαμονής οι οποίες ισχύουν μόνο για τη χώρα μέλος η οποία το εκδίδει και δεν μπορούν να μεταβούν σε καμία άλλη χώρα και δεν μπορούν να επιστρέψουν ε, μέσω διέλευσης από τρίτη χώρα στην χώρα καταγωγής τους. Οποιοδήποτε λοιπόν διαμένει θα πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα σε αυτό το χώρο όπου δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν το κράτος μέλος να σεβαστεί την ελεύθερη κυκλοφορία για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στις περισσότερες χώρες μέλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, οι θεωρήσεις ε, C, D που επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία για τρεις μήνες. Οι θεωρήσεις αυτές θα καταργηθούν από τον Απρίλιο του 2010 όταν θα ε, ξεκινήσει η ισχύ του κώδικα θεωρήσεων. Είναι λοιπόν επίγον να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα και όπως και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει αποφανθεί, πρέπει να συνεχίσουμε την σε αυτού του προβλήματος χωρίς να μειωθεί το επίπεδο ασφαλείας του χώρου Σέγγεν. Πρέπει το σύστημα πληροφόρηση του χώρου Σέγγεν να βελτιωθεί και για τι χώρε έκδοση των ε, θεωρήσεων πρέπει να προβλεφθεί πανομοιότυπη διαδικασία με αυτέ που ισχύουν στι τρίτε χώρε για τι θεωρήσει μακρά διαρκεία. Έτσι λοιπόν θα ανταποκριθούμε στι απαιτήσει ασφαλεία. Επίση, τα κράτη-μέλη πρέπει, εφόσον προβλέπουν θεωρήσει μακρά διαρκεία, να έχουν οπωσδήποτε προηγουμένω βουλευτεί το σύστημα ΣΥΣ, το σύστημα πληροφόρηση, για να είμαστε βέβαια για το επίπεδο ασφαλεία του χώρου Σέγγεν και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα. Όταν κάποια άτομα είναι καταχωρημένα στο σύστημα ΣΥΣ, οι πληροφορίες εφόσον ε, οι υπεύθυνοι τη συμβουλεύονται αποφεύγουμε προβλήματα για τους συνοριοφύλακες ε, στα σύνορα του Σέγγεν. Και βλέπουμε κατά πόσον θεωρήσεις δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να έχουν εκδοθεί, δεν θα πρέπει να τους δοθούν καν. Οι θεωρήσεις μακράς διαρκείας πρέπει να επιτρέπουν ε, την ελεύθερη κυκλοφορία σε τρεις μήνες ή έξι μήνες, ακριβώς με τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για την διαμονή. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δουν κατά πόσον υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό μπορεί να επιτραπεί ως διάστημα για περισσότερο από ένα χρόνο. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Με την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ισχύει νέα νομική βάση για τα θέματα αυτά των θεωρήσεων και βέβαια πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων επί Ισπανικής και Σουηδικής Προεδρίας. Και αυτό εγκαίρως ε, μαζί με τη θέση σε ισχύ του κώδικα των θεωρήσεων. Η Προεδρία της Ισπανίας θα πρέπει να εγγυηθεί στο Κοινοβούλιο αυτό ότι ο κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 5 Απριλίου του 2010. Είναι καθοριστική σημασία ο στόχος αυτός να επιδιωχθεί κατά τρόπο ώστε να αποφύγουμε το νομικό κενό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίκαιρα, λοιπόν, σωστά και έγκαιρα έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία μετά τις ενέργειες της Σουηδικής και Ισπανικής ε, Προεδρίας και εδώ ευχαριστούμε και την σκόδη συγητή της Επιτροπής Λίμπε για τις ε, για το έργο του και την έκθεση που ετοίμασε. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνοντα το επίπεδο ασφαλεία του χώρου Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπο κύριε Μάστρομ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όπως είπε ο εισηγητή, στόχο είναι η κυκλοφορία προσώπων τρίτων ε, υπηκών τρίτων χωρών κατόχων θεώρηση μακράς διάρκειας. Σύμφωνα με το σημερινό κεκτημένο του Σέγγεν, μπορούν ε, τα πρόσωπα αυτά να κυκλοφορούν ελεύθερα, διότι άδεια διαμονής τους ε, ισοδυναμεί με θεώρηση διαβατηρίου. Ωστόσο, πρόσφατα τα κράτη-μέλη έχουν την τάση να μην μετατρέπουν τις ε, θεωρήσεις μακράς διάρκειας σε άδεια διαμονής. Γι' αυτό και το συζητούμε σήμερα, διότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να βρουν μια λύση στο πρόβλημα η νομική και η πρακτική κατάσταση έχει σημαντικές επιπτώσεις για ε, πολίτες τρίτων χωρών ε, που διαμένουν ε, νόμιμα στα κράτη μας. Δεν μπορούν να ταξιδεύουν ούτε να περνούν καν από την επικράτεια μιας χώρας μέλους αν θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και το παράλογο της υπόθεσης στοιχειοθετείται από το παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Κόεγιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη δεν εκδίδουν ε, τις άδειες που ε, πρέπει, τις άδειες διαμονής εν καιρός. Γι' αυτό καταθέτουμε την πρόταση αυτή έτσι ώστε η αρχή της, της ε, αντιστοιχίας μάλλον να επεκταθεί και σε θεωρήσεις μακράς διαρκείας. Χωρίς να χρειάζεται λοιπόν άδεια διαμονής κάποιος, ε, θα μπορεί να ταξιδεύει ε, ε, επί ένα τρίμηνο με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους σαν να είχε άδεια διαμονής. Και είναι και η φιλοσοφία αυτή που διέπει τη δημιουργία ενός εσωτερικού χώρου χωρίς σύνορα να μπορεί ο κάτοχος μιας τέτοιας βίζας μακράς διάρκειας να ταξιδεύει. Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι ο κύριος Κάλλος Κουέιο προτείνει να υποστηριχθεί η πρόταση αυτή από την αρχή μάλιστα και σε συνεργασία με την Επιτροπή νομικών υποθέσεων η Επιτροπή Ελευθεριών κατάλαβε ότι πρέπει να ληφθεί κάποια δράση για να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών των τρίτων ε, κρατών γιατί εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε εκείνους που διαμένουν νόμιμα ε, στις χώρες μας να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ευχαριστώ τον συγητή για την επικοδομητική του πρόταση. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι πρέπει να βρούμε λύση γρήγορα ειδικά για τον κώδικα θεωρήσεων που ε, στις 5 Απριλίου θα ε, αναθεωρηθεί και θα καταργηθεί ένα ενδιάμεσο καθεστώς θεωρήσεων ε, που ήταν μια προσωρινή λύση. Ελπίζω να ικανοποιηθούν όλα τα μέλη από την τελική πρόταση ε, διότι το συμβαστικό κείμενο εγκρίθηκε από όλα τα θεσμικά όργανα. Για να διασκεδάσω κάποιες ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, σε ό,τι αφορά ας πούμε, την ασφάλεια, έχουμε τροποποιήσει αρκετά το αρχικό κείμενο. Μερικά παραδείγματα, Πρόεδρε. η περίοδος ε, διαρκείας συντομεύεται, θα είναι ετήσια και ε, στη συνέχεια είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να εκδίδουν ε, άδεια διαμονής. Επίσης, συστηματική έλεγχη στο σύστημα ΣΥΣ, του ΣΕΝΓΕΝ. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει συστηματικά να κάνουν ελέγχους στο σύστημα πληροφόρησης Σέγγεν, για να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση για τη ε, βίζα ε, τύπου D. Σε ό,τι αφορά τα βιομετρικά στοιχεία, βεβαίω και αυτό είναι σημαντικό για κάποια κράτη-μέλη, έχει επισυναυθεί, όπω γνωρίζετε, στο σχέδιο κανονισμού πολιτική δήλωση, με την οποία καλεί, Ευρω... καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα βιομετρικών στοιχείων ταυτοποίηση ε, σε σχέση με τις θεωρήσεις αυτές και θα σας ε, υποβάλουμε μέχρι τις 21 Ιουλίου τις προτάσεις μας και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επίσης, το δέχτηκε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθεί ως υποχρέωση στο σχέδιο κανονισμού. Και τέλος, για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των εγγύσεων για την ψηλή προστασία των δεδομένων που απασχολεί το Κοινοβούλιο και το ανησυχεί. Επίσης συμφωνήσαμε σε κοινή δήλωση και καλή ε, το Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τις αντίστοιχες προτάσεις για τη σύμβαση του Σέγγεν ε, σε περίπτωση που υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές καθυστερήσεις μετά το 2012 για το σύστημα ΣΥΣ2. Νομίζω λοιπόν ότι η λύση είναι ισόρροπη, καλά σχεδιασμένη για να προστατεύει και να βοηθάει τους πολίτες των χωρών που διαμένουν νόμιμα, επαναλαμβάνω, στι χώρες μας και ανταποκρίνεται και στη φιλοσοφία μιας Ευρώπης χωρίς εσωτερικά σύνορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή Ελευθεριών, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και τον εισηγητή για την τόσο επικοδομητική του στάση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Η κυρία Βίκστρομ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συνεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αφορά και τις αξίες μας και τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εμπόδια και θα πρέπει να πω ότι όλοι όσοι διαμένουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βλέπουν θετικά αυτό. Αλλά το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για όσους σκοπεύουν να έρθουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά μας είπε ο κύριος Κοέγιου, Οι θεωρήσεις μακράς διαμονής επιτρέπουν ε, στον κάτοχο να μείνει στη χώρα στην οποία έχει εκδώσει την ε, θεώρηση αυτή. Να σας δώσω όμως ένα παράδειγμα. Για τη Σουηδία κάποιος ο οποίος μένει στην Ουψάλα δεν θα μπορεί να πάει στο Παρίσι γιατί δεν έχει θεώρηση για τη Γαλλία και ένας φοιτητή από την Κίνα για παράδειγμα δεν μπορεί να φύγει στη διάρκεια των διακοπών και να πάει σε κάποια άλλη χώρα. Επομένως, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Και ε, η πρόταση αυτή είναι ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα εντός της ζώνης Σέγγεν να μπορεί κάποιος να παραμείνει, σε, να, μένει σε, να διαμένει σε μια χώρα αλλά να μπορεί να μεταβεί και σε άλλες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά, έλαβε υπόψη του και όλα όσα ε, είχα εξετάσει εγώ στη ε, διάρκεια της εργασίας μου για την έκθεση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον μιας θετικής πρότασης που θα αποτελέσει μια ακόμα συνεισφορά προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτε τρίτων χωρών να διαμένουν και να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ακριβώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα χώρο στον οποίο θα πρέπει, είμαστε περήφανοι που θα μένουμε. Έχουμε τώρα μιλητέ από τις πολιτικές ομάδες. Η Κίνγκα Γκάλ για το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, καλωσορίζω την ευκαιρία αυτή που έχουμε να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία πολιτών τρίτων χωρών εντός της επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή σκοπό έχει να διευκολύνει τους κατόχους των θεωρήσεων D, ε, θεωρήσεις μακράς διαρκείας δηλαδή, που είναι συνήθως υπήκοοι τριτών χωρών, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να ταξιδέψουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δώσει μια λύση σε καταστάσεις όπου κάποια κράτη-μέλη, για τον ένα τον άλλο λόγο, δεν είναι σε θέση ή δεν έχουν τη διάθεση να δώσουν άδεια παραμονής στους κατοίκους, στους υπηκόους τρίτων χωρών έχουν τους δικούς τους λόγους και δεν εφαρμόζουν το πλαίσιο Σέγγεν σε πολλές περιπτώσεις. Είναι λοιπόν πολύ καλή κίνηση να προσπαθούμε τώρα να εξέρουμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ιδίω για την κατάσταση όπου οι πίκοοι τρίτων χωρών προσπαθούν να περάσουν σε μια άλλη χώρα και αυτό μοιάζει με ένα προσπέλαστο χειρό κάποιες φορές ως προσπάθεια. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή διαχείριση στα θέματα αυτά λοιπόν. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προσπελάσιμα και να αφήνουν τη δυνατότητα να περάσουν οι ταξιδιώτες. Οι υπήκοοι γειτονικών χωρών και εδώ σκέφτομαι ιδίω ουγγρικέ μειονότητε, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν χωρί υπέρμετρο διοικητικό άκτο και δυσκολίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό απαιτείται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών να έχουμε αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα τα οποία να μην αλληλοκαταργούνται αλλά να ενισχύουν από κοινού τους ε, στόχους που έχουμε. Και βεβαίω, κατά πρώτον, θέλουμε να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των φοιτητών, των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν από τέτοιου είδου νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Θα συμφωνήσω λοιπόν ότι η Επιτροπή ω προ το θέμα αυτό θα πρέπει να υποβάλει μία έκθεση μέχρι τον Απρίλιο του 2012, ε, το αργότερο, για την επιβολή του κανονισμού και επίσης ε, να συγκεντρώσει και συμπεράσματα για την εφαρμογή αυτής της, ε, αυτών των διατάξεων. Η κυρία Μπλικεβιτσιούτα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο, για την έκθεσή του. Συμφωνώ απολύτω ότι είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι διασφαλίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκών τρίτων χωρών που βρίσκονται παρόντε στην επικράτεια των κρατών μελών με μια θεώρηση μακρά διαμονή. Ε, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές το να αντικαταστήσουμε την, άδεια, την θεώρηση μακράς διαμονής με μια άδεια παραμονής ε, για υπηκόους τρίτων χωρών είναι μια διαδικασία χρονοφόρα για πολλούς λόγους. Θα μπορούσα να δώσω πολλά παραδείγματα από πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου χώρας, της Λιθουανίας, όπου για παράδειγμα όταν ε, ένας οδηγός με θεώρηση D ε, ένας οδηγός ε, φορτηγού πρέπει να περάσει από το ένα κράτο στο άλλο, πολλέ φορέ δυσκολεύεται να φέρει πέρα στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Έτσι λοιπόν έχουμε επικόστη των χωρών που δουλεύουν ή σπουδάζουν σε κράτη της Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λάβουμε μέτρα προκειμένου οι διαδικασίε έκδοσης θεωρήσεων να απλοποιηθούν για αυτού. Θα πρέπει η ισχύ των θεωρήσεων να είναι η ίδια για την κυκλοφορία των ατόμων εντό του χώρου του Σέγγεν όπως μια άδεια παραμονής. Επίσης, εδώ μια σημαντική πτυχή είναι όχι μόνο η περίοδος ε, της μετακίνησης, του ταξιδιού, την οποία, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο κάτοχος της θεώρησης μακράς διαρκείας, αλλά πρέπει να του δώσουμε και τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες του. Συμφωνώ με την πρόταση ότι οι πίκο τρίτων χωρών που διαθέτουν ε, θεώρηση μακράς διαρκείας σε ένα κράτο μέλο, θα έπρεπε να μπορούν εντό τριών μηνών, ε, μέσα σε οποιοδήποτε εξάμεινο, να μπορούν να ταξιδέψουν σε ένα άλλο κράτο ε, μέλο με τι ίδιε προποθέσει που ισχύουν για του κατόχου των ε, αδειών παραμονή. Η απλοποιημένη μετακίνηση και κυκλοφορία των υπηκών τρίτων χωρών εντό του χώρου Σέγγεν δεν θα έπρεπε να θεωρούμε ότι απειλεί την ασφάλεια των κρατών μελών. Σα απευθύνω λοιπόν έκκληση να εγκρίνετε αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσμπεκ. Eh Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία Επίτροπη. Ακούσαμε ότι υπάρχουν πολλέ δυσκολίε, αλλά ήδη διαμορφώνεται μια διαδικασία με διάφορε φάσει. Και αυτό το κείμενο πολύ καλά μα παρουσίασαν και ε, οι συνάδελφοι, άσχετα από την παράταξη από την οποία προέρχονται, ε, αλλά και ο εισηγητή, είναι μια έκθεση που αφορά όλου του υπηκόου των χωρών που διαμένουν νομίμω στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να εγκριθεί ένα τέτοιο κείμενο και για να εξασφαλίσουμε στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση την ελευθερία των, ε, την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να συμβάλλουμε με ένα ακόμη κομμάτι στο οικοδόμημα τη ε, ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και τη ασφάλεια του χώρου Σέγγεν. Δεν υπάρχουν σοβαρέ διαφωνίε από το κείμενο όπω είδαμε. Και οι περισσότερε τροπολογίε δείχνουν ότι έχουμε όλη τη διάθεση να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που κανεί δεν θα βρίσκεται περιορισμένο σε ένα κράτο μέλο μόνο και θα μπορεί να ανακαλύψει την ε, υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για του υπηκόου, του σπουδαστέ, του ερευνητέ, οποιονδήποτε ζει και εργάζεται στην επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν θα ωφεληθεί και η προεξωτερική προβολή της ε, ε, Ένωσης ως ενιαίου, ως ε, χώρου ενωμένου και θα διασφαλίσουμε, θα προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή πνευματική παράδοση εκτός των συνόρων μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ταβαρές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο, για την πρότασή του. Καθώς και τους και εισηγητές της Επιτροπής Λίμπε. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να πούμε εδώ ότι χρειάζεται να διευκολύνουμε την μετακίνηση των ε, υπηκών τρίτων χωρών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και των τρίτων χωρών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, βεβαίω. Και εδώ βλέπουμε ότι χιλιάδες ε, πολίτες τρίτων χωρών ούτω ή άλλω, συμβάλλουν στην οικοδόμηση αυτού του ευρωπαϊκού χώρου, διαμένουν εδώ, έρχονται για μακρά χρονικά διαστήματα να εργαστούν ή να σπουδάσουν. Συνάδελφοι, λοιπόν, με τη συμβολή του κ. Κοέλιου και των σκεδών εισηγητών, είδαμε πώ μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίε για να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Εδώ ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνο. Ο χρόνο, εφόσον έχουμε να κάνουμε με την ε, καθημερινή ζωή πραγματικών ανθρώπων. Ε, θα μπορούσα να δώσω αρκετά παραδείγματα φοιτητών, ερευνητών, επιστημόνων που φτάνουν στην Ευρώπη γιατί αναγνωρίζεται η εργασία τους ως εργασία ποιότητα αλλά αντιμετωπίζουν κάποιες φορές δυσκολίες ερχόμενοι από άλλες υπήρους γνωρίζουμε ότι κάποιοι ερχόμενοι στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ένα ερευνητή που βρίσκεται στην Πορτογαλία και πρέπει να περάσει στην Ισπανία, βρίσκεται περιορισμένο και δεν μπορεί να ολοκληρώσει λόγω χάρη το μάστερ του για σκοπού έρευνα ή άλλου επιστημονικού σκοπού. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα και είχαμε και άλλε ευκαιρίε. Ε, να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα και γίναν τέτοιες συζητήσεις και στην Επιτροπή μας στην ε, Βρυξέλλες ήδη. Εδώ δεν θέλουμε βεβαίω να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε την κινητικότητα αυτού του είδου των ε, αλλοδαπών ε, πολιτών. Είτε έρχονται από την Κίνα, είτε από την Ινδία, είτε από τη Βραζιλία. Δεν θέλουμε να χάσουμε τι δυνατότητε κινητικότητα του δικού μα του εργατικού δυναμικού, τη επιστημονική κοινότητα και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η αυξημένη κινητικότητα σε περιόδου όπω αυτή που διανύουμε να ενισχυθεί. Και δεν θέλουμε βεβαίω να πληγεί και η κοινωνία τη γνώση. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή το Συμβούλιο να υλοποιήσει αυτέ τι προτάσει προτού τον Απρίλιο τεθεί σε ισχύ ο κώδικα των θεωρήσεων και δημιουργήσει περισσότερου φραγμού και δυσκολίε για την ελεύθερη μετακίνηση των ελευθερών πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν και από τη δική μα την ομάδα στηρίζουμε την, την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα ο κύριο Μπάτεν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση λέει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να δίνουν θεωρίες μακράς διαμονής για ε, διάρκεια 12 μηνών για υπηκός τρίτων χωρών που αναγνωρίζ... και θα αναγνωρίζονται από χώρες μελή της Σέγγεν. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στη Σέγγεν, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις, αλλά οι προτάσεις αυτές θα διευκολύνουν τους πολίτες ε, χωρών μελών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να μεταβούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η Βρετανία έχει τεράστιο πρόβλημα με την παράνομη μετανάστευση. Έχουμε ε, εκατομμύρια ε, παρανόμως διαμένοντες στην Βρετανία και ουσιαστικά αυτοί που διαμένουν στην Βρετανία παρανόμως θα μπορούν να έρθουν σε μια άλλη χώρα μέλος ε, με νόμιμο τρόπο, παραδείγματο χάρη στη Γαλλία και από εκεί και πέρα να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως το UKIP θα καταψηφίσει αυτή την πρόταση για να μην ε, βοηθήσει, μη συνδράμει περαιτέρω στην παράνομη μετανάστευση. Ευχαριστώ κύριο Φανχέκε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην έκθεση διαβάζω ένα περίεργο λόγο γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε την περίπτωση. Ας πούμε ένας ξένος φοιτητής ε, που ε, σπουδάζει στο Βέλγιο και μετά θέλει να πάει σε μια βιβλιοθήκη ε, στη Ολλανδία και μετά ταξίδι στη Βαρκελόνη. Ωραίο είναι για το φοιτητή, καλά περνάει. Αυτό είναι όμως το Σέγγεν, αυτή είναι η πρακτική. Ο στόχος δεν είναι να ταξιδεύουν ελεύθερα οι φοιτητέ, να, να ανοίξουμε διάπλατα τα σύνορα για ε, τη λαθρομετανάστευση, για το δουλεμπόριο. Και δεν υπάρχουν σύνορα όπως στο, παρελθόν ε, ήταν πυλώνας η προστασία των σύνορων. Είδαμε στην Ισπανία πώς έγινε μαζική ε, νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών που μπορούν τώρα ελεύθερα να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ να σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για τους ε, Ευρωπαίους και να μην σκέφτεστε την καθημερινή ε, δουλειά και τα ταξιδάκια των ξένων φοιτητών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα Γαρσία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον καλό Κοέγιο για την εξαιρετική του δουλειά και κυρίω για το υψηλό επίπεδο συνένεση που πέτυχε με το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διάφορα ε, κόμματα, και πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο. Ε, λίγα είναι τα σημεία που διαφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το μεγαλύτερο χώρο ελευθερίας που είναι γνωστός. Θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα εμπόδια που παρεμποδίζουν ελεύθερη κυκλοφορία και για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση. Έχουμε παράλογες καταστάσεις. Συχνά αντιμετωπίζουν εκείνοι που έχουν ε, ε, θεωρήσεις μακράς διαμονής και θα πρέ... τύπου ΔΕΛΤΑ και θα πρέπει να τερματιστούν αυτές οι καταστάσεις. Όπως γνωρίζετε, οι ε, θεωρήσεις αυτές επιτρέπουν στους κατόχους να ε, διαμένουν στη χώρα που τους έχει χορηγήσει τη θεώρηση. Ωστόσο δεν μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν στην Ένωση εκτός ε, όταν επιστρέφουν στη χώρα που ε, έδωσε αυτή τη θεώρηση. Πολύ συχνά λοιπόν βλέπουμε καταστάσεις όπως περιγράφηκα. Να σας δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα. Κάποιος κάνει διδακτορικό στη Λισαβόνα για την ιστορία της Αμερικής και ε, δεν μπορεί να πάει στη Σεβίλη που απέχει μία ώρα με το αεροπλάνο ε, στο ε, αρχείο των Ινδιών το λεγόμενο για την ιστορία της Λατινικής Αμερικής να προετοιμάσει το διδακτορικό του. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να διευκολύνουμε την αρχή της κυκλοφορίας, ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους κυρίως εργασιακούς και επιστημονικούς και σπουδών. Τέλος, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, ε, τους οποίους εκτιμώ και σέβονται, να υποστηρίξουν την έκθεση του κυρίου Κοέλιο, που είναι εξαιρετικής ποιότητας και όχι μόνο. Είναι και εγγύηση, ακόμα μια εγγύηση υπέρ της μεγάλης ε, ε, ελευθερίας, χώρου ελευθερίας και ε, διέλευσης. Ευχαριστώ Κάρλος, την Ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιατόβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο, για το έργο του και για την συνεργασία που είχε μαζί μα, αλλά και με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την ε, κατάρτιση τη έκθεση αυτή. Ελπίζουμε ότι η ανάγνωση αυτή θα είναι και η τελευταία. Είναι καθοριστική σημασία πριν το τέλο του Απριλίου 2010 να εγκριθεί η έκθεση αυτή, ώστε να τεθεί σε ισχύ ε, και να εγκριθούν αυτέ οι προτάσει μαζί με τον κώδικα θεωρήσεων. Είναι σημαντικό όλα τα άτομα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ταξιδέψουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίω δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί από την ε, ισχύ των θεωρήσεων ε, στην περίπτωση που δεν ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για τι άδειε παραμονή. Θα πρέπει λοιπόν ένα άνθρωπο που έχει θεώρηση μακρά διαρκεία να μπορεί να ταξιδέψει παντού στην Ευρώπη και να μπορεί ο υπεύθυνο επίση να λάβει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε όταν εκδίδει την θεώρηση και να πληροφορείται κατά πόσον η θεώρηση αυτή αυτομάτω μπορεί να μετατραπεί σε άδεια παραμονή πριν την εκπνοή του πρώτου χρόνου ισχύω. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε το γεγονό ότι για λόγου ασφαλεία κάθε άτομο που θέτει υποψηφιότητα για να λάβει θεώρηση D θα πρέπει να επαληθεύεται αν ε, περιλαμβάνεται στο σύστημα SIS ή όχι, το σύστημα πληροφόρηση των θεωρήσεων. Είναι σημαντικό οι πληροφορίε που περιλαμβάνονται στο ΣΥΣ να παρέχονται αγκαίρω σε όλου του συμβαλωμένου στο σύστημα αυτό. Το σύστημα ΣΥΣ 2 ούτω ή άλλω δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλο του 2012. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλουν τι απαραίτητε νομοθετικέ προτάσει για να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο προστασία όπω και αυτό που είχαμε μέχρι τώρα από το ΣΥΣ. Ευχαριστώ κύριο Μποργέτσιο για ένα λεπτό. Αυτές οι προτάσεις θέλουν να διευκολύνουν τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν μονή, νόμιμα σε μία χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, ε, το χώρο Σέγγενς και την ελεύθερη μετακίνηση χάρη στη θεώρηση τύπου D. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να επεκτείνουμε αυτή τη δυνατότητα και να υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ άδεια παραμονή και θεώρηση ε, μακρά διαρκεία τύπου D. Ουσιαστικά θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με την άδεια παραμονή για την ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο Σέγγεν. Με άλλα λόγια, θέλουμε να επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε κατέχει ένα έγγραφο νόμιμη διαμονή να κυκλοφορεί ελεύθερα στο χώρο Σέγγεν για σύντομε περιόδου, οι οποίε δεν υπερβαίνουν του τρει μήνε. Ε, και εμείς θέλουμε να καταγγείλουμε αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Είναι ήδη ε, πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τα πράγματα σε μια τρίτη χώρα και καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι ελοχεύουν με την ε, σαφή εφαρμογή αυτής της αρχής. Ευχαριστώ κύριο Σόμπερ Μάιερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγου μήνε, χαιρόμασταν, ήταν και Χριστούγεννα και ε, πολλοί συνάδελφοι χάρηκαν γιατί χαλάρωσε το σύστημα της θεώρησης. Μαυροβούνη, Μακεδονία, ε, Σερβία ε, και τα λοιπά και έχουμε ένα κύμα μέσω της ε, Αυστρίας μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες. 150.000 περίπου Μακεδόνες ζήτησαν ε, και έκαναν χρήση αυτής της ρύθμισης ε, ο μιλητής. Και δύο στους τρεις δεν γυρίζουν πίσω. Είναι ολόκληρη μετανάστευση λαών, μετακίνηση. Πέντε λεωφορεία την ημέρα να βλώνουν από τη Μακεδονία για τη Βόρεια Ευρώπη. Βέβαια είναι τουρίστες αυτοί και απαγορεύεται να εργαστούν. Τι σημαίνουν όλα αυτά μετά από 90 μέρες βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Υποτιθέμενοι τουρίστες ε, δουλεύουν ε, σε τιμές dumping και στην παράνομη οικονομία. Ιδού λοιπόν η ε, διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις χήμερες και τα όνειρα που ζουν εδώ ορισμένοι. Και ποιος τα υφίσταται όλα αυτά, τα κράτη-μέλη, οι πατρίδες μας. Αυτό που ψηφίζει εδώ η πλειοψηφία. και έχουμε παράνομη μετανάστευση και μαύρη εργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούσουτιλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Κάρλος Κοέλιο για την έκθεσή του και για αυτή την πρωτοβουλία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να υποφεληθούν της ελευθερίας μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επισημάνω ένα στοιχείο ηρωνίας που έχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Παρά το γεγονός ότι δίνουμε άδεια ουσιαστικά σε υπηκόους τρίτων χωρών, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα για τις δυνατότητες τους να ταξιδέψουν από χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρε όπω η Λιβύη, για παράδειγμα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την Ελβετία και τη Λιβύη. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η Λιβύη δεν εκδίδει θεωρήσεις ε, σε πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο σε Ελβετούς πολίτε. Επομένω, εμεί έχουμε λιγότερο, μικρότερα, λιγότερα δικαιώματα να ταξιδεύουμε σε τρίτε χώρε, όπω για παράδειγμα η Λιβύη. Οι συνέπειε είναι πολύ σοβαρέ, διότι έχουμε εργαζομένου που δεν μπορούν να μεταβούν για να εργαστούν στη Λιβύη, έχουμε επιχειρήσει που δεν μπορούν να αποστείλουν του εργαζομένου του, ε, όπω επίση και επενδυτέ και έχουμε και εργαζομένους που βρίσκονται στη Λιβύη και πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι να αποσταλεί ο αντικαταστάτης τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση και θα ήθελα να ζητήσω από την Επίτροπο Γόλστρομ να δράσει καταπηγόντως για το θέμα αυτό ε, καταλαβαίνω ότι είναι διπλωματικό θέμα μεταξύ δύο χωρών που δεν είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι συνέπειες είναι σοβαρές και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα αυτή για να μπορέσουν να κερδίσουν τα προστοζήν. Ευχαριστώ. Η Μόνικα Φλασίκοβα Μπένοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση του κ. Κοέλιο και η πρόταση για κανονισμό αφορούν ένα κεντρικό στοιχείο τη δημοκρατία στην Ευρώπη, δηλαδή την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Είναι απαράδεκτο οι κάτοχοι ε, θεώρηση μακρά διαρκεία για μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να λάβουμε τέτοιε πρωτοβουλίε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σεβαστούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ακριβώ την ελεύθερη μετακίνηση. Εάν ένα κράτο μέλο επιτρέπει σε έναν υπήκοο τρίτη χώρα να παραμείνει στην επικράτειά του, δεν υπάρχει κανένα λόγο το άτομο αυτό να μην μπορεί να μετακινηθεί σε ολόκληρο το χώρο του Σέγγεν. Προφανώ πρέπει να επεξεργαστούμε με προσοχή τι λεπτομέρειε, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο προστασία και ασφάλεια στο χώρο Σέγγεν δεν θα μειωθεί. Όμω, Νομίζω ότι στην ε, ομάδα των ανθρώπων κατά των οποίων ασκούμε διακριτική μεταχείριση, όπω του φοιτητέ ε, και του ερευνητέ, θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτού και του επιχειρηματίε, οι οποίοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε ο κύριο Μπορή για το έλεγχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κοέλιο. Έχω ασχοληθεί και εγώ με την έκθεση αυτή και τον κανονισμό. Η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο επίγουσα, είναι και συμβολική. Και μπορώ με περηφάνεια να πω ότι σήμερα ως εκπρόσωπος ενός νέου κράτους μέλους βοηθάω να αλλάξει νομοθεσία για να διευκολύνεται η κυκλοφορία ε, πολιτών ε, στο χώρο Σέγγεν. Μέχρι πρόσφατα οι χώρες μας ε, γνώριζαν τις ίδιες δυσκολίες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύτιμη η συμβολική σημασία της ε, απόφασης αυτής. Η κατάργηση των ε, θεωρήσεων ε, C και D και η αδυναμία των κρατών να εκδίδουν άδειες παραμονής προκαλούν πολλά προβλήματα. Άλλο παράδειγμα, ένα ζευγάρι Ουκρανών φοιτητών που τους σταμάτησαν στα σύνορα γιατί δεν εγνώριζαν ε, την κατάσταση. Ε, ήταν φοιτητές, ήθελαν να πάνε κάπου για να ενημερωθούν για τις σπουδές τους και τους συνέλαβαν. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε το σύστημα ανταλλαγής προφοριών του Σέγγεν ΣΥΣ 2 και να βελτιώνουμε την ομοθεσία μας. Καλό με λοιπόν την κυρία Επίτροπο να φροντίζει να είναι καλύτερος ο συντονισμός αν όχι τόσο καλό όσο τώρα. Ευχαριστώ η κυρία Γκιόνις επόμενη. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή και Υποστηρίζω την έκθεσή του, υποστηρίζω όμω και την κυρία Μάλμστρομ. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσει και την ασφάλεια. Ξέρω ότι πολλά ζητάω, ε, θα περιοριστώ σε λίγα όμω. Για να ε, λειτουργήσει σωστά ο κανονισμό αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε πρώτα απ' όλα και να γνωρίζουμε περισσότερα για τι πρακτικέ που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα κράτη δίνουν ε, άδειε παραμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι καλές οι πρακτικές και αυτές θα πρέπει να τις αναλύσουμε και να τις εναρμονίσουμε για να υπάρχει και μεγαλύτερη ε, αλληλο εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Όλοι μιλούν για το σύστημα ΣΥΣ, ε, δεν το χρησιμοποιούν όλοι όμως και καλό θα είναι να ενταχθεί το σύστημα ΣΥΣ 2 το συντομότερο, να γίνει μετάβαση από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2, να λειτουργεί σωστά και είναι προς ε, όφελος και συμφέρον της Ευρώπης οι πολίτες τρίτων χωρών να λειτουργούν σωστά και να κυκλοφορούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ καταρχάς τον κύριο Κοέλιο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει για αυτή την έκθεση και να πω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, το κεκτημένο της συνθήκης Σέγγεν συνιστά ακριβώς αυτό, την ελεύθερη κυκλοφορία εντός των ορίων ε, του, της περιοχής Σέγγεν επομένως στην συζήτηση αυτή πρέπει να βγάλουμε το πρώτο βασικό και απλό συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτός ο κανονισμός και ε, το παράδειγμα του φοιτητή είναι χαρακτηριστικό όποιος έχει θεώρηση μακράς διαμονής να έχει το δικαίωμα ε, ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας. τίθεται η προβληματική και σε αυτό θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή κατά πόσο θα ε, διευκολυνθεί έστω και με τρόπο έμεσο η παράνομη μετανάστευση αν θα υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας ή κατά πόσο ε, κάποιος ε, εφαρμόζοντας αυτό το δικαίωμα δεν θα μπορεί να ε, έχει παράλληλα και τα μέσα για να κινηθεί και επομένως τα κράτη μέλη θα έπρεπε να το λαμβάνουν αυτό υπόψη. είναι δεδομένο ότι κάθε κράτος μέλος όταν εκδίδει τις θεωρήσεις πάντα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό και στο σημείο αυτό τίθεται μια πολύ σημαντική παράμετρος όπως ορίζεται στην έκθεση που είναι η πλέον καθοριστική ότι στο σύστημα πληροφοριών σέγγεν πλέον θα είναι υποχρεωτική η ε, επεξεργασία των δεδομένων πριν τη θεώρηση μακράς διαμονής. άρα τελικά όχι μόνο διασφαλίζουμε το κεκτημένο τη συνθήκη σέγγεν τελικά ενισχύουμε και την ασφάλεια ε, σε ό,τι αφορά ε, αυτό ακριβώς το δεδομένο και ως εκ τούτου όλοι πρέπει να είμαστε ε, θετική στην προοπτική αυτή και βεβαίως σε κάθε περίπτωση γρήγορα να προχωρήσει το σύστημα sis ii που είναι απαραίτητο και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες των κρατών μελών όχι μόνο να διευκολύνουμε το κεκτημένο σέγγεν και να το ενισχύσουμε να ενισχύσουμε παράλληλα και την ασφάλεια που είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε κράτος μέλος για όλους μας για το κεκτημένο της συνθήκης αυτής. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Next speaker Στη συνέχεια η Τάνια Φαϊόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι η άρση των συνόρων και η διασφάλιση της ελεύθερης μετακίνησης ε, προσώπων. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα στον χώρο Σέγγεν. Ορισμένε φορέ λόγω γραφειοκρατία δεν επιτρέπουμε σε φοιτητέ, ερευνητέ αλλά και σε άλλου να κινούνται ελεύθερα. Κυρίω πολίτε τη Σερβία, του Κωσυφοπεδίου, οι οποίοι παραδόξω έχουν λιγότερα δικαιώματα από όσα απολάμβαναν στο παρελθόν. δεν θα πρέπει να υποκύπτουμε σε δεδομένα που δίνουν ε, ε, τεράστια στοιχεία για παράνομη μετανάστευση ε, να μας κάνουν να μην επιτρέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν ελεύθερα ορισμένες φορές κάνουν αίτηση για θεωρήσεις και αυτές απορρίπτονται ακριβώς λόγω των στοιχείων της παράνομης μετανάστευσης. Η ίδια διάκριση γίνεται και σε νέους, οι οποίοι ορισμένες φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την Ευρώπη. Υπάρχει η Αλβανία, η Βοσνία, η Ριζεγοβίνη, οι οποίοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένου όρους για την ε, απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και όλο αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα προς τα μπρο και θα είναι φυσικά και προς το συμφέρον τη Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση που έχουμε αφορά μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άρση των συνόρων και η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει της προσοχής μας. Η παρούσα κατάσταση είναι παράλογη και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο άτομα τα οποία κατέχουν θεωρήσεις μακράς διαρκεία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο χώρο της Έγγεν, ενώ άτομα τα οποία έχουν θεωρήσει μικρής διάρκειας μπορούν. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκής επιτροπή είναι καλή, αλλά χρειαζόμαστε και κάποιε δικλείδε ασφαλεία, όπω ακριβώ πρότεινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. αυτοί που βρίσκονται στον ε, κατάλογο μη αποδεκτών προσώπων του ΣΥΣ ε, θα πρέπει ε, να κοινοποιούνται και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και υποστηρίζω και την προθεσμία της 5ης Απριλίου του 2010. Υποστηρίζω την πρόταση σε γενικές γραμμές. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch Η κυρία Λουκασεύσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το Σέγγεν και η ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Πιο εύκολα κυκλοφορούν εκείνοι που έχουν θεώρηση ε, βραχιάς διάρκειας από εκείνους που έχουν θεώρηση μακράς διάρκειας. Κάποιο που διαμένει ε, νόμιμα και μόνιμα στην Πολωνία δεν μπορεί να φύγει να πάει στη Γερμανία ταξίδι. Και μιλήσαμε για τους ερευνητές, για τους επιστήμονες, για τους φοιτητές, για τους επιχειρηματίες. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, να επισκεφτούν τους φίλους τους, να γνωρίσουν τις παραδόσεις, τις χώρες και να γίνουν καλοί πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστρέφοντας τις χώρες τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόλτσερ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα βίζα των χωρών Σέγγεν είναι από ό,τι φαίνεται τόσο περίπλοκο που δεν ξέρουν πια οι προξενικοί υπάλληλοι τι να κάνουν και πώς να δίνουν ε, τις θεωρήσεις. Είναι και παγίδα οι θεωρήσεις. Κατηγορίες D και C ε, είναι ε, επίσης κάτι που δεν γνωρίζουν ε, οι υπάλληλοι των προξενείων και δίνουν τις βίζες εκείνες που είναι πιο εύκολο να δοθούν και δεν χρειάζεται να συμβουλευτούν το σύστημα ΣΥΣ. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα αυτά και δεν χρησιμοποιείται καν το σύστημα προειδοποίησης του ΣΥΣ. Τώρα τι συζητάτε για εθνικά συστήματα και δράπεζες δεδομένων. Ε, βλέπουμε να αυξάνονται οι αιτήσει ασύλου και, και τώρα ε, επαπειλείται κύμα μεταναστεύσεως από τα Βαλκάνια πάνω περίπου 150.000 πολίτες της Μακεδονίας ε, σειραίουν προς την Κεντρική Ευρώπη και δεν γυρίζουν πίσω, ιδίω στους τρεις είπαμε. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Ευχαριστώ κυρία Μόρβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς οι Ούγγροι εκπρόσωποι ε, έχουμε περίεργη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να αποφασίζουμε με τη ψήφο μας για το εάν θα διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτών τρίτων χωρών ή αν ε, θέλουμε να την περιορίσουμε αυτή την ελεύθερη ε, κυκλοφορία. Η Ουγγαρία μετά από τη τραγωδία του Τριανού έχασε πολύ ε, μεγάλο τμήμα της επικράτειάς της και έχουμε πολλούς αδελφούς Ούγγρους οι οποίοι ζουν εκτός των σημερινών συνόρων της Ουγγαρίας και εκτός των σημερινών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι αδελφοί μας, οι Ούγγροι, ε, ζουν μια κατάσταση ταπείνωσης κάθε φορά. έρχονται και σπουδάζουν, ε, εργάζονται και ε, κάνουν ερευνητικό έργο στην σημερινή ακροτηριασμένη Ουγγαρία που είναι η πατρίδα τους και μετά δεν μπορούν να πάνε πουθενά άλλου. Είναι πολύ κακή η κατάσταση, αφόρητη θα τη χαρακτήριζα και θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε. Γι' αυτό εμείς οι Ούγγροι βουλευτές θα ε, ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόντς. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή βασίζεται στην εικασία ότι όλοι οι πολίτε των τρίτων χωρών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλόπιστοι. Και αν λένε ότι έρχονται εδώ για να σπουδάσουν, αυτό πραγματικά και κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω έχει και ψευδοκολέγια τα οποία φαίνεται να έχουν καταλόγου με φοιτητέ, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν εμφανιστεί σε ένα μάθημα. Κάποιοι λοιπόν, εφόσον διευκολυνθεί η μετακίνησή του σε άλλα κράτη-μέλη, θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν ω προ το αν πραγματικά σπουδάζουν, για το κατά πόσο το καθεστώ του είναι αληθινό. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται βέβαια, δεν συμμετέχει στο χώρο Σέγγεν, ε, όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματικά ρυθμού ρεκόρ για την ε, νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Οι σημερινοί κάτοχοι θεωρήσεων μακρά διαρκεία και αδειών παραμονή μπορεί να είναι οι παράνομοι μετανάστε του αύριο και οι ελεύθεροι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μετακινούνται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόν. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μάλστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Δύο ερωτήματα κυρίω τέθηκαν, όχι ακριβώ σχετισμένα με αυτήν την έκθεση, αλλά θα ήθελα σύντομα να τα θίξω. Ο κύριος Μπουζούτιλ μίλησε για τη Λιβύη. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα ε, και βεβαίω είμαστε σε ενεργό διάλογο με τη Λιβύη και με την Ελβετία και με τα άλλα κράτη-μέλη προκειμένου να αναζητήσουμε μια κατάλληλη λύση στο πρόβλημα αυτό πριν υπάρξει κλιμάκωση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να επανέλθω και να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις. Τον κύριο Φαγιάν να πω ότι βεβαίω η κατάσταση τη Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια άλλη περίπτωση, ξεχωριστή. Θέλουμε να οριστικοποιήσουμε την εξέταση τη κατάστασή του για να δούμε κατά πόσον οι χώρε αυτέ ανταποκρίνονται στα κριτήρια. Η Επιτροπή, η Επιτροπή έχει ήδη διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη και ετοιμάζει έκθεση για το θέμα αυτό. Η αξιολόγηση ε, είναι κάτι που θα σα παρουσιάσουμε εν ευθέτω χρόνο και ενδεχομένω να υποβάλουμε και μια σχετική πρόταση και να τη συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξή μα. Τώρα, για την ε, προκειμένη πρόταση, να διαβεβαιώσω του ε, βουλευτέ και τον εισηγητή ότι πραγματικά έχουμε σκοπό το έργο αυτό να το προωθήσουμε και να βεβαιωθούμε ότι οι διατάξει αυτέ θα υλοποιηθούν. Μπορεί να φαίνεται το πρόβλημα να είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά δεν είναι. Αφορά συγκεκριμένου πολίτε, συγκεκριμένα άτομα και θέλουμε να ενθαρρύνουμε του ανθρώπου να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίμω. Ερευνητέ, ε, σπουδαστέ, επιστήμονε, φοιτητέ, γιατί είναι καλό και για εκείνου και για και βεβαίω αυτή είναι και η φιλοσοφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε δηλαδή έναν χώρο ε, χωρί εσωτερικά σύνορα. Θέλουμε λοιπόν να μην γίνει ακόμη πιο περίπλοκη η ζωή των ανθρώπων αυτών. Με την πρόταση αυτή λοιπόν νομίζω έχουμε ξέβρει μια σωστή ισορροπία. Και Νομίζω ότι λάβαμε υπόψη και τι ανησυχίε περί ασφαλεία κατά ικανοποιητικό τρόπο και ε, ενώ νομίζω ότι οι τρεις, τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάστηκαν και συνεργάστηκαν με άριστο τρόπο. Αναζητήσαμε σε συγκεκριμένα προβλήματα χειροπιαστές λύσεις προκειμένου να ωφελήσουμε τους πολίτες. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Κοέλιο για το έργο σας και ευχαριστούμε για αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση στην Ολομέλη. Thank Ευχαριστώ κύριε Επιτροπή. και τέλος ο εισηγητής μας ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τέσσερα πολύ σύντομα, τέσσερις σύντομες σημειώσεις πρώτα απ' όλα. Λυπάμαι που στο θέση του Συμβουλίου δεν κάθεται κανεί κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρομ για τη συμπαθητικά τη λόγια και για τη βοήθεια που μα έδειξε, καθώ και τη βοήθεια του Συμβουλίου βεβαίω. Θα πρέπει να, να να φροντίσουν για την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού εντό τη 5η Απριλίου. Και γιατί αλλιώς θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για ανθρώπους, πραγματικούς ανθρώπους. Έπειτα, να εκπρέσω την γιατί υπήρξαν ε, συνάδελφοι που θύμισαν τα προβλήματα ασφαλείας, αλλά δεν αναγνωρίζουν οι συνάδελφοι αυτοί ότι το Κοινοβούλιο βελτίωσε τον κανονισμό με τις προτάσεις του. Κυρίως την υποχρέωση της πρώτερης ε, εξέτασης του τι συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, του ΣΥΣ. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και ενισχύει την ελεύθερη κινητικότητα αλλά και την ασφάλεια που θέλουμε να διασφαλίσουμε στο χώρο Σέγγεν. Αρκεί να δει κανεί. Ε, το θέμα είναι να μην βλέπει κανεί ένα μέρο τη αλήθεια, αλλά το σύνολο, ολόκληρη την αλήθεια. Και τέταρτον, ε, Πρόεδρε, ήθελα να, να ευχαριστήσω όσου συνεργάστηκαν για να επιτύχουμε το στόχο μα και τους ε, υπευθύνου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και όλου, από όλε τι πολιτικέ ομάδε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, οι οποίοι φρόντισαν να δημιουργηθεί αυτή η συνενετική εξέταση του θέματος. Ελπίζω λοιπόν ότι το πρόβλημα με την προσπάθειά μα αυτή θα λυθεί και ότι βέβαια δείχνουμε ότι κάνουμε την δουλειά μα κατά τον πλέον άριστο τρόπο. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Πέρας λοιπόν της συζήτησης, η ψηφοφορία θα γίνει τόσο λίγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να παραμείνετε στην αίθουσα ή να πάτε έξω μια βόλτα. Διακόπτουμε μέχρι τις 12 η ώρα. Ευχαριστώ.